Colleagues, please take your seats. Αδελφοί, καθίστε. Παρακαλώ, να ξεκινήσουμε. Please take your seats. Παρακαλώ, καθίστε. σε γεγό και τα λοιπά. Okay. Okay, I'll make a start. Please take a seat also the λοιπόν, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ καθίστε και οι κύριοι εδώ στην πρώτη σειρά. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ καθίστε. Και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ηρεμήστε, θα συνεχίσετε μετά. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού, με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να προεδρεύσω προσωρινά μέχρι να εκλέξουμε πρόεδρο. Δεν είμαι ο πρεσβύτερος ε, ευτυχώς, αλλά είμαι ο παλαιότερος ευρωβουλευτής, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και ελπίζω να μην μοιάζω και γυριότερος μετά τη συνεδρίαση. Λοιπόν, άρχεται η συνεδρίαση. Διερμηνία υπάρχει σε όλες τις επίσημες γλώσσες, ε, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Προεδρείου. Να σας υπενθυμίσω ότι σκοπός αυτής της συνεδρίασης είναι να συσταθεί σε σώμα το Προεδρείο της Επιτροπής με την εκλογή Προέδρου και τεσσάρων αντιπροέδρων σύμφωνα με το άρθρο 213 του κανονισμού. Θα εκλέξουμε πρώτα Πρόεδρο και μετά Αντιπροέδρους υπό την Προεδρία του νέου εκλεγέντος ε, Πρόεδρου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με ειδοποιούν ότι συμμετέχουν οι εξής αναπληρώτες... Α, και άλλη αλλαγή, μάλιστα. Από το ΕΛΚ. Ο Βλαντιμίρ Μπίλτσικ αντικαθιστά τον κύριο Μπερλοσκόνη. Αντρέι Αλίσκι αντικαθιστά την Σάντρα Καλνιέτε. Χαβιέρ Σαρσαλέχος αντικαθιστά την κυρία Σουίτσα. Ο κύριος Ανδρίου Κουμπιλίους θα γίνει τακτικό μέλος ε, στη θέση της ε, κυρίας Μπέντελε. Η σχετική επιστολή εστάλει στις 8 Ιουλίου. Από τους ο κύριος Ατίλα Αράκοβατς αντικαθιστά τον κύριο Ανδρέα Σίντερ. Ο κύριος Ρούπερτ Χάιζελ αντικαθιστά την Κάτι Πύρη από τους πράσινους. Η Χάνα αντικαθιστά την Σαλή Γένμπου. Από το κόμμα ID ο Νικόλας Μπέι αντικαθιστά τον Χάραλτ Βιλίμσκι. Από το ECR ο Σίτο Κάνκο αντικαθιστά την Άννα Ο κύριος Άνχελ Τζαμπάσκι αντικαθιστά τον Κάρολ Κάρσκι και ο Μπέρτ Γιάν Ρόισεν αντικαθιστά τον κύριο Βάιμελς. Και από τους μη εγγεγραμμένους ο Μύροσλαβ Ραντατσόφσκι αντικαθιστά τον κύριο Λάντς Φόρμαν και επιπλέον από την άλλη ο Φρεντερικ Ρίς ή Φρεντερικ Ρίς αντικαθιστά τον Μπερνάρ Κέστα. Αυτοί είναι οι αναπληρωτές. Αν υπάρχουν και άλλες αλλαγές, μπορούν οι πολιτικές ομάδες να ενημερώσουν ε, τον πρόεδρο τώρα, αλλά νομίζω ότι ε, έχουν ειδοποίησει για όλες τις αλλαγές. Τέλος, πριν ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω ε, να φροντίσετε να έχετε όλοι τις κάρτες για την ψηφοφορία, αυτές εδώ. Μπορεί να τις χρειαστείτε στην διαδικασία. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι όλοι οι υποψήφοι πρέπει να δεχτούν ε, αυτοπροσώπως ή γραπτός ε, την υποψηφιότητα πριν από οποιαδήποτε εκλογή και πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής και να έχουν υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και την δήλωση που αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 213 παραγραφός 1, αναφέρω κατά λέξη η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην σύνθεση του Προεδρείου κάθε επιτροπής. Δεν θα επιτρέπεται να υπάρχει ένα Προεδρείο μόνο με άνδρες ή μόνο με γυναίκες ή όλοι οι αντιπρόεδροι να είναι από την ίδια χώρα μέλος. Οπότε, περνάμε τώρα στο σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, εκλογή Προέδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω από την γραμματεία να διαπιστώσει ότι έχουμε απαρτία. Με ενημερώνουν ότι έχουμε απαρτία. Υπάρχουν σίγουρα 38 τακτικά μέλη. Να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 218 η απαρτία είναι 1 τέταρτο των μελών. Στην περίπτωσή μας 18, εφόσον έχουμε 38 έχουμε σίγουρα απαρτία. Θα ήθελα τώρα να ε, ζητήσω υποψηφιότητες ε, για την θέση του Πρόεδρου. Κυρία Ζόφκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Ντέιβιντ Μακάλιστερ για Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ. Έχουμε μία υποψηφιότητα λοιπόν του κυρίου Ντέιβιντ Μακάλιστερ. Να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να προταθεί από πολιτική ομάδα ή από 5% των μελών της Επιτροπής, δηλαδή τέσσερις βουλευτές. Ε, προκειμένου, προτείνεται από μια πολιτική ομάδα. Ο κύριος Μακάλιστερ ε, δέχεται την υποψηφιότητα. Βλέπω μου κάνει νόημα. Ο υποψήφιος ε, είναι και τακτικό μέλος της Επιτροπής. Έχει υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και την δήλωση για τον κώδικα συμπεριφοράς. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Μια που υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, σας ζητώ να εκλεγεί διαβοής. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αρκεί. Ε, εκλέγαμε και άλλους με τόσο χειροκρότημα. Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο να αναλάβει. Εμένα τελείωσαν τα καθηκοντά μου. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας ε, σε μένα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που θα συνεχίσω να προεδρεύω των εργασιών της ΑΦΕΤ για άλλα δυόμιση χρόνια. Θα προσπαθήσω να προεδρεύω όσο πιο αμερόληπτα μπορώ και όσοι συνάδελφοι ήσαν εδώ κατά την προηγούμενη θητεία θα γνωρίζουν ότι έχω βέβαια το προσωπικό μου στυλ αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο δίκαιος γίνεται για όλα τα άτομα, όλε τι πολιτικές ομάδες, Ούτω ή άλλω δεν είναι καθήκον του Προέδρου να δρά με προκατηλημένο τρόπο. Και για όσους ε, μόλις ε, εξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μέλη τη Επιτροπή μα, σα συγχαίρω για την εκλογή σα, σα συγχαίρω που είστε μέλη αυτή τη Επιτροπής, γιατί αντικειμενικά από όλε τι 20 επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή η επιτροπή είναι η καλύτερη και η πιο ελκυστική. Συμφωνούμε έτσι, δεν είναι. Νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουν όλε οι άλλε 19 επιτροπέ. Εδώ είναι οι καλύτεροι. Να συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία μα. Ευχαριστώ πολύ τον Μίχαελ Γκάλα για την ε, εναρκτήρια διαδικασία. Σημείο 2. Εκλογέ αντιπροέδρων. Λοιπόν, θα έχουμε ε, διαδοχικές, χωριστές ε, εκλογές. Ενημερώθηκα ότι η εξή αναπληρωματική συμμετέχω στην ψηφοφορία. Να το ξαναδιαβάσω. Όχι, ωραία, ευτυχώς. Οπότε, λοιπόν, υποψηφιότητες για τον πρώτο αντιπρόεδρο. Ο κύριος Σάρος Βόλσκι. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι και πάλι στην ΑΦΕΤ. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Από πλευράς της ομάδας ECR θέλω να προτείνω για, ως πρώτο αντιπρόεδρο της ΑΦΕΤ, τον κύριο Βαστσικόφσκι, εδώ αριστερά μου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνικής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάτσεκ Σαρισβόλσκι, υπενθυμίζω ότι πρέπει να προταθεί ο υποψήφιος από μια πολιτική ομάδα από 5%. Οπότε το ECR προτείνει τον κύριο Βασκόφσκι ως πρώτο αντιπρόεδρο. Τώρα θέλει να μιλήσει ο κύριο Πίτσουλα από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Συγχαρητήρια. Από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θέλω να προτείνω για τρίτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής τον κύριο Σέργεϊ Στάνισεφ. Πρώτο ή τρίτο. Τρίτο. Τρίτο. Τρίτο. Τρία. Ε, ε, Τονίνο, in the moment we're still... Τονίνο, ε, είμαστε όμως ακόμη στην εκλογή του πρώτου αντιπρόεδρου. Λοιπόν, κύριε Βασικόφσκι, συμφωνείτε με την υποψηφιότητά σας. Ναι. Οπότε, είναι τακτικό μέλος, έχει υπογράψει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και ε, και σωστής συμπεριφοράς. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Χίλτε Βάουτμανς, από τους φιλελεύθερους, από το, συγγνώμη, το Ρινιού. Το Κοιτάξτε, δεν έχω συνηθίσει ακόμη. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε στην προηγούμενη θητεία και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σωστά. Τον κύριο μας Πάρτ θέλω να τον ε, προτείνω για δεύτερο αντιπρόεδρο. Α, είμαστε στο... Α, καλά για τον πρώτο αντιπρόεδρο, εμεί ως Renew θέλουμε να υπάρξει μυστική ψηφοφορία για, αυτήν την, ε, για αυτό το διορισμό. Καλώ. Από τη μία. Μάθαμε και για τον τρίτο αντιπρόεδρο, ποιο προτείνεται. Αλλά έχουμε και το αίτημα για μυστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία. Πρέπει να το ζητήσει τουλάχιστον το 1 πέμπτο των μελών δηλαδή 15. Πρέπει να ρωτήσω, ποιοι θα ήθελαν να υπάρξει μυστική ψηφοφορία. Παρακαλώ μετρήστε. Επαρκής. Προφανώς, άνω των 15. Άνω των 15. Και τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Ε, να ψηφίσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, τις κάρτες σας. Λοιπόν, για τους ε, νέους υπάρχουν κάποια κουμπιά εκεί. Πράσινο είναι υπέρ, το κόκκινο είναι κατά. Λευκό είναι αποχή. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για τον διορισμό του κυρίου Βασουκόφσκη ως πρώτου αντιπροέδρου. Μυστική ψηφοφορία. So, has everyone voted? Ψηφίσατε όλοι. Ένα συνάδελφο ακόμη δεν έχει ψηφίσει. 66 από του 67, παρακαλώ. Όχι εγώ, όχι εγώ. Τώρα όμω έχουμε ένα παραπάνω. Όχι, 68 παρόντε. Ε, ε, ε, ψήφισαν και 68 πέρα. Και όταν αποτέλεσμα. 37 υπέρ, 24 ε, κατά. Συγχαρητήρια κύριε Βασκόφσκι. Οπότε, τρίτο σημείο. Λοιπόν, υποψηφιότητε για τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αντιπρόεδρο. Οι σοσιαλδημοκράτε, από ό,τι ξέρουμε, λοιπόν. πάει για Ρινιού για δεύτερο αντιπρόεδρο. Τρίτο αντιπρόεδρο Στάνισεφ, σοσιαλιστής. Και για την τέταρτη. Από πλευρά του ΕΛΚ προτείνω τον κύριο Μπασέσκου. Ωραία. Συμφωνούν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουμε. Παγιέτ, Στάνισεφ και κύριο Παζέσκου. Και οι τρεις συμφωνούν, αλλά έχουμε την εξής κατάσταση. Όπως ξέρετε, το άρθρο 2.13 λέει, για να ε, αντανακλάτε η διαφορετικότητα του Κοινοβουλίου στο Προεδρείο κάθε Επιτροπή δεν επιτρέπεται να είναι το Προεδρείο αποκλειστικά να αποτελείται από άνδρες ή από γυναίκες και είτε όλοι να είναι από το ίδιο κράτος μέλος. Προφανώς όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι ε, προτάθηκαν δεν είναι από το ίδιο κράτος μέλος, αλλά είναι όλοι άνδρες. Άρα, για να σεβαστούμε τους κανόνες, η έκθεση, αλλιώς η εκλογή του Προεδρείου θα ακυρωθεί όλων των μελών του Προεδρείου. Γι' αυτό δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα αλλά να αναβάλω την εκλογή των επόμενων αντιπροέδρων για να επιτρέψω στις ομάδες να εξετάσουν την υποβολή άλλων υποψηφιότητων. Όπως σας υπενθυμίζω, ούτως ή άλλως μετά την εκλογή του Προέδρου και του πρώτου αντιπροέδρου έχει συσταθεί κανονικά σε σώμα και μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί η Επιτροπή μας, αλλά έχουμε αυτή τη δυσχέρεια. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ένα Προεδρείο που να αποτελείται μόνο από άντρε. Τώρα κάποιοι έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μπίτιχοφ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε απόλυτος υπέρ της απόφασής σας να αναβάλουμε, διότι πρέπει να δοθεί ίση ευκαιρία σε όλες τις πολιτικές ομάδες να επανεξετάσουν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Πίτσουλα. Κύριε Πρόεδρε. Εξετάζοντας βεβαίως αυτό που είπατε, πρέπει καθότι είναι τεχνικά δυνατό να μην αναβάλουμε την ψηφοφορία μέχρι και τον τρίτο αντιπρόεδρο προκειμένου να επιτύχουμε την απαραίτητη ισορροπία φύλου. Πρόεδρος, η κυρία Βιλανουέβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Κύριε Πρόεδρε υποστηρίζομαι την αποφασή σας να αναβληθεί η εκλογή, διότι μιλούμε για την διεύθυνση πρόεδρο και αντιπροέδρος για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι θεμελιώδης για το μέλλον του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό για το πρόσωπο που έχουμε με τους συνομιλητές μας, είναι απαράδεκτο να μην έχουμε ούτε μία γυναίκα υποψήφιο και να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να είναι αυτό η πρώτη μας απόφαση. Χωρίς να εκπροσωπούμε δηλαδή το ίμιση του πληθυσμού και στις διευθυντικές ομάδες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Γκάλα για το ΕΛΚ παρακαλώ. Ναι Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με την αναβολή έχουμε κάποιες αντιφατικές διατάξεις στους κανόνες για το Κοινοβούλιο αφενό και αφετέρου την ελευθερία των πολιτικών ομάδων να προτείνουν τα ονόματα που θεωρούν κατάλληλα, τα μέλη που θεωρούν κατάλληλα. Και στην περίπτωσή μας και νομίζω και σε δυο τρει άλλε επιτροπέ οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και επομένως δεν εξαρτάται από εμά αυτή τη στιγμή να εξαντλήσουμε Δηλαδή να εκλέξουμε δεύτερο και τρίτο αλλά όχι τέταρτο αντιπρόεδρο δεν θα ήταν δίκαιο. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να ξαναδούν το θέμα και άρα πράγματι πρέπει να διακόψουμε την περαιτέρω συγκρότηση σήμερα. Μάλιστα κύριε Γκάλα. Ε, κύριε Φάκου ε, ίσως ε, έπρεπε να δούμε την ε, κατάσταση αυτή προτού ψηφίσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο. Γνωρίζω ότι προχωρούμε με τον πρόεδρο και πρώτο αντιπρόεδρο, αλλά είχαμε τις υποψηφιότητες. Δηλαδή θα ήθελα να δώσω και στο ECR να δώσουμε τη δυνατότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα γυναίκας. Σας ευχαριστώ, λέει πρόεδρος όλες οι πολιτικές ομάδες προφανώς έχουν ικανές γυναίκες συναδέλφους και το ΕΛΚ και άλλοι. Γιάτσεκ, ε, πρόεδρε, ήθελα απλώ να πω ότι έγινε αυτό. Αν είναι να ακολουθήσουμε την πρόταση του Ρινιού, θα πρέπει να ακυρώσουμε την εκλογή του πρώτο αντιπροεδρού, το οποίο δεν θα ήταν το σωστό. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρος, είναι μια δύσκολη κατάσταση, ελπίζω να την είχαμε αποφύγει. Δεν κατέστη δυνατό, αλλά ο κανονισμός είναι τόσο σαφής που είμαστε υποχρεωμένοι. Ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι να διατηρήσουμε τα πράγματα ως έχουν με τον κύριο Βασικόφσκι πρώτο αντιπρόεδρο, να καθίσουμε με τις ομάδες και να βρούμε μια λύση. Για να συμμορφωθούμε προς το άρθρο 2.13. Δεν βλέπω άλλη δυνατότητα. Άκουσα από τους σοσιαλιστές ότι θέλουν να συνεχίσουμε. Όλες οι άλλες ομάδες από ό,τι κατενόησα είναι υπέρ της πρότασής μου να διακόψουμε εδώ τη διαδικασία. Καλά δεν τα λέω. Επ' αυτού πρέπει να ψηφίσουμε, δεν νομίζω. Είναι σαφέ. Επομένω, ανακοινώσει τώρα από τον πρόεδρο το επόμενο σημείο, σύμφωνα με το 2.14, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει αρμοδιότητε για λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων στους συντονιστές, με εξαίρεση την έγκριση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων και τροπολογιών. Κάθε πολιτική ομάδα εκπροσωπείται στους συντονιστές και οι μη εγγεγραμμένοι ενημερώνονται μέσω των ε, συμβούλων τους. Αν δεν έχουμε αντιρρήσεις, θεωρώ ότι αυτό εγκρίνεται, η απόφαση αυτή εγκρίνεται, ωραία. Τώρα, έχετε λάβει το χρονοδιάγραμμα, το ημερολόγιο του υπολείπου για το έτος, αν δεν έχω αντιρρήσεις και αυτό θεωρώ ότι έχουμε εγκρίνει, Το γλωσσικό τώρα προφίλ της Εντροπής ΑΦΕΤ, σύμφωνα με τα μέλη της και προηγούμενες αποφάσεις Προεδρίου, καλύπτονται 20 γλώσσες. Lithuanian, Latvian, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian and Swedish. If there are no objections... Αν δεν έχετε αντιρρήσεις από πλευρά σας μπορούμε να εγκρίνουμε αυτό το γλωσσικό καθεστώς, λέει ο Πρόεδρος. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι έκτακτη Τετάρτη 24 Ιουλίου 9 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι. Το σχέδιο διατάξεως θα σας αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτά από μου. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία τα επόμενα πέντε χρόνια.